You know, I cannot stand this. Τσακ, τσακ, τσακ. Καλησπέρα. Τι χαρά που σας βλέπω. Καλύτερα όμως να καθίσετε για να αρχίσουμε. And I would advise you all for, for the coming meeting. Και τις επόμενες φορές να έρχεστε στην ώρα σας. Είναι καλύτερα να αρχίζουμε στις 3 και όχι στις 3 και 4. Πράγματα είναι αυτά. Πρέπει βέβαια να είναι κανείς Πολωνός για να εκτιμάει την τάξη φαίνεται. Σας κατευχαριστώ λοιπόν. Σας καλωσορίζω. Θα περάσουμε καλά σήμερα. Όπως ξέρετε έχουμε τρεις μισοήμερες συνεδριάσεις και παρακαλώ να είστε υπομονετικοί γιατί εγώ έχω πολύ μεγάλο κρύαμα και δεν ακούω ούτε τι λέω. Αν δείτε ότι φωνάζω να μου το πείτε και αν δείτε ότι μιλάω πολύ χαμηλόφωνα να μου το πείτε και αυτό. Αλλά έχω μεγάλο συνάχη. Με μεγάλη χαρά και τιμή καλωσορίζουμε εδώ και αναφέροντες εκπροσώπους κρατών μελών και εκπροσώπους της Κομισιόν. Για τα πρακτικά, για τις αναφορές που θα συζητήσουμε σε αυτή τη συνεδρίασή μας, θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω ότι για την αναφορά 344 κάθετος 14 για αύριο θα, θα εξεταστεί μαζί με μια άλλη γιατί έχει το ίδιο θέμα. Και επίσης υπάρχει αίτημα να ξανανοίξει η αναφορά 1660 που θα τη βρείτε στην προσθήκη των σημειωμάτων της Προεδρίας. Είναι μια Ιρλανδική αναφορά για την χρηματοπιστωτική κρίση. Δεν είμαι πλήρως πεπισμένη ότι θα ήταν λογικό και σωστό να ξανανοίξει αυτή η αναφορά, διότι δεν έχω πιστεί ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι για να προχωρήσει. Αλλά επειδή είναι σημαντικό θέμα και αξίζει την προσοχή μας, θα έλεγα να το προωθήσουμε στους συντονιστάς για πλήρη συζήτηση και απόφαση. Αν συμφωνείτε κι εσείς, νομίζω ότι είναι ευρύ το θέμα και πρέπει να το συζητήσουμε παραπάνω από ό,τι θα μπορούσαμε τώρα. Εντάξει, ωραία, ευχαριστώ πολύ. Τώρα, το σημαντικότερο θέμα που έχω να σας πω σήμερα είναι να προσέξουμε όλοι και οι συνάδελφοι και το προσωπικό και όλοι ότι ο προϊστάμενος της γραμματείας μας ο David Lowe φεύγει στη σύνταξη στο τέλος του μήνα και θα έχουμε την ευκαιρία να γιορτάσουμε την αποχώρησή του και την καριέρα του και θα οργανωθεί μια δεξίωση στο τέλος της αυριανής συνεδρίασης το βράδυ εδώ απ' έξω. Παρακαλώ να έρθετε και να του πείτε οτιδήποτε θέλετε, είναι έτοιμος για όλα. Επίσης μπορώ να σας ανακοινώσω σήμερα την παρουσία της κυρίας Βίρπλη Πούπα που έχει οριστεί νέα επικεφαλής της γραμματείας μας από την 1η Φεβρουαρίου. Σηκωθείτε μια στιγμούλα Η Βίλπε έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Είναι Φινλανδή και τα περασμένα πέντε χρόνια ήταν επικεφαλής της υπηρεσίας του Ιντρανέτ. όχι μόνο του Κοινοβουλίου και άλλων Ιντρανέτ και άλλων εργαλείων για εσωτερική επικοινωνία. Και ήταν επικεφαλής 35 ατόμων. Προηγουμένως ήταν διοικητική υπάλληλο στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, στην Υπηρεσία Τύπου κλπ. Και ακόμη πριν ήταν ερευνήτρια στο Φιλανδικό Υπουργείο Εργασίας. Χαιρόμαστε λοιπόν ιδιαίτερα για την παρουσία σου σήμερα και προσβλέπουμε σε στενή και αποτελεσματική συνεργασία. Επίσης μπορώ να σας αποκαλύψω ότι μιλάει τέλεια σου ειδικά. Γι' αυτό να προσέχετε. Να προσέχετε. Α, όχι αστεία το λέω. Μιλάει πολύ καλά σου ειδικά λοιπόν. Και έτσι θα μάθω και εγώ μαζί της μερικά φιλανδικά. My Αυτά είχα να σας πω. Και τώρα Κάτι άλλο ενδιαφέρον. Mr. Ambroise Ο κύριος Πέχαρ είναι εδώ. He left the room obviously, but he is ο Πολωνός σύμβουλος για τους σοσιαλιστές και αυτός φεύγει στη σύνταξη. Α, και αυτός φεύγει. Αλλά δεν θα φύγει τελείως θα γράψει ένα βιβλίο για τους σοσιαλιστάς στο κοινοβούλιο από το 79 και μετά. Θα τον βλέπετε για αρκετό καιρό λοιπόν. Πάντως να του γνωστοποιήσετε ότι το ανακοίνωσα όπως έπρεπε και να τον μεταφέρετε τους χαιρετισμούς μου. Και τώρα το πρόγραμμα να δούμε αν το εγκρίνεται ή αν έχετε καμία αντίρρηση. Μπορούμε να δεχτούμε την ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τίποτε άλλο που θα θέλατε να συζητήσουμε πριν αρχίσουμε. Όχι, πάμε κατευθείαν στις αναφορές. Η πρώτη είναι του Μίχα Ρέγκατσαρ. Εξ ονόματος πολλών υπογραφώντων για την προστασία της περιφέρειας κράση στη Σλοβενία από κερδοσκοπία σχετική με ακίνητη περιουσία και από την καταστροφή μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Βλέπω με χαρά ότι έχουμε εδώ Σλοβαίνους βουλευτάς και τους καλωσορίζω. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν Τόμας Βίντμαν. Εδώ είναι, εδώ είναι. Α, εκεί είναι, από εκεί. Α, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Τόμας Βίτμαν λέγομαι, από τη Γενική Διεύθυνση ΦΙΣΜΑ. Uh, um, Το πρόβλημα με την αναφορά αυτή είναι ότι η διατύπωση δεν ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρη, δεν ήταν πάρα πολύ σαφής και νομίζω ότι ήδη το 2011 δική επιτροπή είχε ασχοληθεί με την αφορά αυτή και από όσο καταλαβαίνω ο αναφέρον ζήτησε στη συνέχεια να δοθούν περισσότερες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να αποσαφινιστεί το ζήτημα. Από όσο γνωρίζουμε όμως εμείς δεν έδωσε περαιτέρω στοιχεία ο ίδιος ο αναφέρον όπως όφιλε. Ωστόσο βλέπουμε ότι ο αναφέρον έχει δύο σημαντικές ανησυχίες. Πρώτον, η προστασία της περιφέρειας Κράς της Σλοβενίας κατά της μόλυνσης του περιβάλλοντος και η δεύτερη ανησυχία που είναι και πιο σημαντική έχει να κάνει με την διασφάλιση του όλου μπορούμε να πούμε γεωργικού περιβάλλοντος, διασφάλιση της απαραίτητης παροχής γεωργικών τροφίμων και γενικότερα διασφάλιση της καλλιέργειας στην περιοχή. Και από ό,τι φαίνεται υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι ξένοι, κυρίως αλλοδαποί, οι οποίοι αγόραζαν μεγάλα κτήματα στην περιοχή Εκράσα. Και κατά αυτόν τον τρόπο αυξήθηκε η τιμή των αγροκτημάτων. Ο αναφέρον όταν υπέβαλε το 2011 για πρώτη φορά την αναφορά αυτή, περίμενε από τη σκοβενική κυβέρνηση να περιορίσει την αγορά ακίνητης περιουσίας, την αγορά γης από τους λοδαπούς. Επί της αρχής όμως αυτό αντιβαίνει στην ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων. Ωστόσο, βλέπετε επίσης από το φάκελό σας ότι μέχρι το Μάιο του 2011 η Σλοβενία καθώς επίσης και άλλες χώρες είχαν τη δυνατότητα να προασπίσουν, να προστατεύσουν για τους δικούς τους ουσιαστικά τους υπηκόους την αγορά γης και μπορούσαν κατά αυτόν τον τρόπο να αποκλείσουν την αγορά γης από λοδαπούς. Ξέρετε ότι αυτό προβλέπεται από τη συνθήκη προσχώρησης για μία περίοδο 7 ετών μετά την προσχώρηση. Το 2011 όταν υποβλήθηκε η αναφορά αυτή, η Σλοβενία είχε τότε τη δυνατότητα να ζητήσει μία επέκταση, μία παράταση για επιπλέον τρία χρόνια αυτής της προθεσμίας, αυτής της δυνατότητας. Και φαίνεται ότι ο αναφέρον αυτή τη στιγμή καταγγέλει το ότι η Σλοβενική κυβέρνηση δεν ζήτησε αυτή την περαιτέρω παράταση. Προφανώ η Σλοβενία δεν είναι υποχρεωμένη να ζητήσει μια τέτοια παράταση, επομένω για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υπάρχει καμία παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Ωστόσο, η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, η βασική δηλαδή αυτή αρχή, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί διακριτική μεταχείριση με βάση την υπηκότητα, την εθνικότητα. Μπορούν όμως να λαμβάνονται μέτρα προκειμένου να αποθαρρυνθούν αγοραστές οι οποίοι αγοράζουν γη για λόγους κερδοσκοπίας ή μπορούν να προβλεφθούν κάποια μέτρα προκειμένου τμήματα γης να διατηρηθούν για την καλλιέργεια, για σκοπούς αγροτικής ανάπτυξης. Δεν λάβαμε πάντως εμείς περαιτέρω στοιχεία από τον αφέροντα και θεωρούμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μπορεί να κλείσει η αναφορά αυτή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε τώρα να κάνουμε συζήτηση με τους συναδέλφους. Ο κύριος Μπόκοβιτς έχει το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως εξήγησε και ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η συγκεκριμένη αναφορά έχει ανοίξει εδώ και κάποια χρόνια στην, και αφορά την περιφέρεια, την περιφέρεια Κράς. Μία περιφέρεια στην οποία βλέπουμε ότι έχει αλλάξει εντελώς το χωροταξικό σχέδιο με διάφορες αποφάσεις που είχε πάρει και η ίδια η κυβέρνηση και έχουμε δει και πάρα πολλές τροποποιήσεις έκτοτε. Στο παρελθόν είχαμε ένα χώρο που υπήρχαν κυρίως αγροκτήματα και μικρά σπίτια και στη συνέχεια είδαμε ότι υπήρχαν πάρα πολλοί αγοραστές και από την ίδια την Σλοβενία αλλά και από την Ιταλία και μια έντονη οικοδομική δραστηριότητα και όλα αυτά τα είδαμε κυρίω μετά την ένταξη τη Σλοβενία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ συμμετείχα τότε στο Κοινοβούλιο τη Σλοβενία και είχαμε υποβάλει ένα ερώτημα προ τον τότε Πρωθυπουργό, ζητώντα να σταματήσει η οικοδομική αυτή δραστηριότητα, η αγορά τη γη και είχαμε ζητήσει περαιτέρω προστασία αυτή τη περιφέρεια, τη περιφέρεια Κρά. Όπω είπατε, όντω η σλοβενική κυβέρνηση δεν έλαβε κάποια συγκεκριμένα μέτρα το 2011 για την προστασία της περιοχής. Ωστόσο αυτό που βλέπουμε είναι ότι η τιμή της γης και κυρίως αγροτικής γης έχει εκτοξευθεί, είναι πολύ ψηλότερη από ό,τι ήταν στο παρελθόν, έχει δεκαπλασιαστεί σε ορισμένες περιπτώσεις και βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πίκοοι της Σλοβενίας οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση πλέον στην αγροτική αυτή γη, δεν μπορούν πλέον να καλλιεργήσουν τη γη Προτείνω λοιπόν το ακόλουθο. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να ζητήσουμε από την κυβέρνηση της Σλοβενίας να αναλάβει εν μη άλλο κάποια δράση για να προστατεύσει την περιφέρεια κράση καθώς επίσης και τους κατοίκους της περιφέρειας αυτής έτσι ώστε να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να έχουν πρόσβαση όντως στην αγροτική γη. Σας είχα πει ότι σχετικό ερώτημα είχα υποβάλει εγώ, καθώς επίσης και η πολιτική μου ομάδα το 2011 στο Σλοβενικό Κοινοβούλιο. Κάποια πράγματα μπορούσαν να γίνουν τότε, η κατάσταση έχει τροποποιηθεί σήμερα, 9 και 2015, μολονότι έχουμε καθυστερήσει, θεωρώ ότι ακόμα και τώρα μπορούμε να λάβουμε μια κάποια δράση. Ο κύριος ευχαριστώ μου δίνετε το λόγο κυρία Πρόεδρε. Όπως ακούστηκε ήδη, η Σλοβενία είχε τη δυνατότητα να εξασφαλίσει προστατευτικά μέτρα μέχρι μία επταετία το πολύ μετά την προσκόρησή της, από την ημερομηνία της ένταξης δηλαδή και μετά. Αλλά δυστυχώς δεν ελήφθησαν ενεργά μέτρα, δεν δραστηριοποιήθηκε τότε η κυβέρνηση της χώρας και οι αρμόδιες αρχές. Εμείς υποστηρίζουμε απολύτως το πνεύμα αυτής της πρωτοβουλίας των πολιτών, αλλά ε, ιδιαίτερα από την περιβαλλοντική του σκοπιά. Και επίσης, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Σλοβενίας, θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη όλες οι πτυχές ε, και οι ε, οπτικές, ας πούμε, της αναφοράς. Βεβαίως, θα πρέπει να συμμορφούνται προς την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία που μεταξύ άλλων εξασφαλίζει την υψηλή προστασία της βιοπικιλότητας και των υδατίνων πόρων και βεβαίως και την πολιτιστική κληρονομιά και γενικότερα τη φύση. Η κυρία Φαγιόν. Δεν θέλω να πω τίποτα. Άλλος κανείς από συναδέλφους, ακόμα και αν δεν είναι Σλοβαίνος, ο κύριος Πέτερ Γιάρ. Καλά, μην σπρώχνεστε. Θέλετε να διαφωνήσετε εκτός της αιθούσης. Ε, ποιος θα μιλήσει πρώτος. Ναι, εκείνος πρώτος λέει ο κύριος Γιάρ και μετά εγώ. Ο κύριος Κύρο, Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Βλέπουμε ότι προκύπτουν τέτοιες καταστάσεις όταν από τη μία πλευρά Έχουμε μία επίσημη αναγνώριση, όπως εδώ πέρα από την UNESCO για την περιοχή αυτή, η οποία πλέον ανήκει στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Και από την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θέλουν τελικά να σφετεριστούν ένα τμήμα της γης αυτής, που επίσημα ανήκει στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Πρέπει λοιπόν σαφώ να αποφύγουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα κερδοσκοπική και θα πρέπει κυρίως να μπορεί να συνεχίσει η περιφέρεια αυτή να νίκει στον κατάλογο μνημείων της UNESCO, γιατί μπορεί η ουσιαστικά να αυτή να αποσυρθεί αν δεν υφίστανται οι απαραίτητες συνθήκες προκειμένου να γνωρίσει την περιφέρεια αυτή ως περιφέρεια παγκόσμιας κληρονομιάς. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά τα στοιχεία. Άκουσα προσεκτικά και τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Θα πρέπει λοιπόν η σλοβενική κυβέρνηση να ανταποκριθεί στην αναφορά αυτή. Θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και να δούμε τελικά αν μπορεί η σλοβενική κυβέρνηση, αν προτίθεται τελικά, να αναλάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσει την περιφέρεια κράση. Νομίζω λοιπόν ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένο να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή, διότι βλέπουμε ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση για το ζήτημα αυτό και κυρίως για την πολύ όμορφη και πολύτιμη αυτή περιφέρεια Κράσα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γιάρ, θέλετε το λόγο. Όχι, με κάλυψε ο συνάδελφος. Λοιπόν, μπορούμε να προτείνουμε τώρα το εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να κλείσουμε την αναφορά, υπάρχουν όμως κάποια θέματα που θέλουμε να διευκρινίσουμε. Όχι ότι θα επηρεάσουμε την κυβέρνηση, τουλάχιστον να πούμε τη γνώμη μας. Θεωρώ λοιπόν ότι οι Σλοβαίνοι συνάδελφοι θα επιθυμούσαν να στείλουμε εμείς επιστολή στην κυβέρνηση και να τους βολιδοσκοπήσουμε για τις προθέσεις τους και τα μελλοντικά τους σχέδια και μέχρι τότε μπορούμε να κλείσουμε την αναφορά. Πάντα καλό είναι όμως να εκφράζει τις απόψεις σου και να πούμε ότι παρακολουθήσαμε το θέμα τουλάχιστον, ασχοληθήκαμε και διαπιστώσαμε ότι νομικά δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να προχωρήσουμε, αλλά τουλάχιστον λέμε τη γνώμη μας. Συμφωνείτε με αυτό, ο κύριος Γιάρ. Συμφωνώ απολύτως με την πρόταση της Προέδρου, αλίμονο, μια μικρή συμπλήρωση μόνο. μπορεί να βοηθάει τους Σλοβαίνους συναδέλφους. Μπορούμε να πούμε ότι ένα μεγάλο τμήμα των προβλημάτων πρέπει να λυθούν στα κράτη-μέλη. Και σε περίπτωση που υπάρχει Επιτροπή Αναφορών στη Σλοβενική Βουλή, πράγμα που δεν γνωρίζω, να συστήσουμε στους πολίτες να αποτείνονται στην Βουλή τους και στην ε, δική τους Επιτροπή Αναφορών, γιατί είναι και πιο άμεσος ο διάλογος. Ως συμπλήρωση για να πούμε στον αναφερόμενο ότι πολλά έχουν να κάνουν με το περιθώριο χειρισμών και λιγμών της ίδιας της χώρας τους και να μην απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δηλαδή, αλλά στην εθνική τους. Βεβαίω με κάποια φιλική διατύπωση, όχι ομά και απότομα, όπως πάντα φιλικά και ευγενικά. I don't think there is a petitions... Δεν νομίζω ότι υπάρχει στη Σλοβενική Βουλή Επιτροπή Αναφορών. Α, υπάρχει! Α, τότε καλά. Ας κάνουμε λοιπόν αυτό, να στείλουμε επιστολή στην κυβέρνηση με αντίγραφο στην Επιτροπή Αναφορών. Ναι, εντάξει, να κλείσω, να κλείσω. Κλείνω. Επόμενη. Η αναφορά για μια απαγόρευση πο, πώλησης πυτεριγίων Καρχαρία στην Ένωση. Α, ναι, Καρχαρία. Πυτεριγίων ο Αλέξανδρος Στάιν από την Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχατε ήδη πάρει μια γραπτή απάντηση από την Κομισιόν και δεν άλλαξε τίποτε από τότε, γι' αυτό θα συνοψίσω σύντομα. Εμείς δεν είμαστε σε θέση να προτείνουμε απαγόρευση της πώλησης πτυρυγίων Καρχαρία, γιατί το υπάρχον νομικό πλαίσιο προβλέπει ότι οποιαδήποτε βιώσιμη συναλλαγή πρέπει να επιτρέπεται. Για την προστασία προστατευομένων ειδών πρέπει να ληφθούν άλλου είδους μέτρα αλλιευτικά. Γι' αυτό εμείς τονίζουμε ότι παίζουμε τον κύριο ρόλο για την προστασία των καριχαριών με διαφορετικούς όμως τρόπους. Πρώτον, απαγορεύεται η αλίευση τους σε ενωσιακά ύδατα και δεύτερον προβλέψαμε μία μεταρρύθ, μία τροπολογία που έκανε πιο αυστηρή την απαγόρευση αυτή από τους Φινλανδούς αλληλείς. Τρίτον, εφαρμόζουμε μέτρα για την απαγόρευση της αποκοπής και, πώλησης, ε, της αποκοπής και αλίευσης πτερυγίων καρχαρία πέρυσι τον Νοέμβριο η Επιτροπή αλληλία του Βορειοανατολικού Ατλαντικού πανέλα αυτή την απαγόρευση αλίευσης των καριχαριών Και τέλος, επίσης προστατεύουμε το είδος του καρχαρία μέσω της εφαρμογής διεθνών συμβάσεων όπως το ΣΑΙΤΕΣ ή τη σύμβαση για τα μεταναστευτικά είδη. Έχουμε μάλιστα συμπεριλάβει και τρία πρόσθετα είδη καρχαριών στα απαγορευόμενα προσαλίαν. Άρα παίζουμε σημαντικό ρόλο για την προστασία του είδους του καρχαρία και επίσης επιτηρούμε, παρακολουθούμε την πρόοδο της εφαρμογής της σύμβασης ΣΑΙΤΕΣ για να δούμε μήπως υπάρχουν μη βιώσιμες συναλλαγές επ' αυτών. Και αν διαπιστωθεί τίποτα τέτοιο θα πάμε στον ΠΟΕ. Ευχαριστούμε πολύ. Άρχεται η συζήτηση. Κόντιλ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα πρέπει να πω ότι δεν είναι αηφόρος η αλία του Καρχαρία. Προφανώς. Αν δούμε ε, τις ε, πηγές που ασχολούνται με αυτά τα θέματα ε, θα διαπιστώσουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός των καρχαριών που αλλιεύονται και φωνεύονται και μάλιστα σε μεγάλα βάθη πέφτουν μέσα σε ε, δίχτυα. Το 1996 ήταν απειλούμενα 15 είδη καρχαρία. Το 2010 αυτά τα είδη έχουν φτάσει στα 80. Ε, έχουμε καταλάβει λοιπόν ότι θα πρέπει κάτι να κάνουμε για αυτή την υπόθεση και να απαγορεύσουμε την ε, αλήψη καρχαρία. Δεν υπάρχει αηφόρος αλία όπως έχουμε σήμερα Κανείς άλλος δεν έχει ζητήσει το λόγο. Αν δεν απατώμε. Προτείνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, αλλά η Επιτροπή Αλίας έχει εγκρίνει μια πάρα πολύ θετική αναφορά ε, και έκθεση συγγνώμη για αυτή την αναφορά από την τελευταία φορά που το συζητήσαμε. Εμείς πρέπει να κλείσουμε την αναφορά, έτσι προτείνεται, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω, αλλά λαμβάνουμε υπόψη για μελλοντικές αναφορές ε, για αυτό το θέμα ε, ότι τίθεται και πάντα μπορούμε να το συζητούμε. Αλλά εν προκειμένου έχει ήδη συζητηθεί και έχει κλείσει. Προτείνω λοιπόν να κλείσουμε την αναφορά. Διαφωνεί κανείς. Συμφωνείτε όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε. Επόμενη αναφορά. Είναι της κυρίας Πατρίτσια Μπαλτζαρίνη σχετικά με την προστασία του φυσικού καταφυγίου Φόντο Τότσε στο Πεδεμόντιο της Ιταλίας. Και θα δώσω μέσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Μάρκο Σιπριάνη. Thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην αναφορά αυτή η αναφέρουσα καταγγέλει ένα συγκεκριμένο έργο δημιουργίας ενός γηπέδου γκόλφα σε ένα φυσικό καταφύγιο στην περιοχή Πιεμόντε της Ιταλίας. Το φυσικό αυτό καταφύγιο ανήκει επίσης, ε, είναι προστατευόμενος τόπος Natura 2000 όσον αφορά τους οικοτόπους για τα πτηνά. Σύμφωνα λοιπόν με τα αναφέρουσα, η δημιουργία ενός γηπέδου γκόλφα θα υπονόμευε τη φυσική ομορφιά, τη φυσική αξία αυτού του φυσικού καταφυγίου η ε, οδηγία όσον αφορά τους οικότοπους και όσον αφορά τα, την προστασία των πτηνών δεν απαγορεύει την δημιουργία, την κατασκευή οικοδομημάτων στα πλαίσια του Natura 2000. Λέει παρόλα αυτά στα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να κάνουν μια κατά αξιολόγηση του προβλεπόμενου έργου προκειμένου να δούνε αν το έργο αυτό θα μπορούσε τελικά να έχει σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά τον λόγο φυσικό καταφύγιο. Επομένως, θα πρέπει να γίνει μια μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων σε κάθε περίπτωση. Αν τώρα το πόρισμα της εκτίμησης αυτής είναι αρνητικό, τότε το έργο αυτό, το σχέδιο αυτό μπορεί να εγκριθεί μόνο σε πολύ συγκεκριμένε περιπτώσεις προβλέπονται από τις οδηγίες, δηλαδή σε περιπτώσεις σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, αν δηλαδή δεν μπορεί να προβλεφθεί καμία άλλη εναλλακτική λύση και αν έχουν προβλεφθεί τα μέτρα αποζημίωσης, αντισταθμιστικά μέτρα. Στα πλαίσια της αναφοράς βλέπουμε ότι υπάρχει και μία τεχνική έκθεση από, την από τον Περιφερειακό Οργανισμό για την Προστασία του Περιβάλλοντος της Περιφέρειας του Πιεμόντε. Ο οργανισμός αυτός εξέτασε μία μελέτη εκτίμηση των επιπτώσεων που έκανε ο ανάδοχος και εντόπισε κάποιες αδυναμίες στα πλαίσια αυτής της μελέτης. Και ο Περιφερειακός αυτός οργανισμός λοιπόν εντόπισε στη συνέχεια κάποια κάποιες ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει το έργο αυτό αν εγκριθεί και τελικά ελοποιηθεί. Βάσει όλων των διαθέσεων πληροφοριών είδαμε ότι οι Ιταλικές αρχές δεν έχουν ακόμα εγκρίνει το έργο αυτό. Επομένως δεν υπάρχει καμία τελική απόφαση εκ μέρους των Ιταλικών αρχών ότι πρόκειται όντως να ελοποιηθεί αυτό το έργο. Συνεπώς, το άρθρο 6.3 της Οδηγίας για τους Οικοτόπους όσον αφορά δηλαδή αυτή την εκτίμηση των επιπτώσεων, βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Επί του παρόντος λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για παράβαση της ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τις Ιταλικές Αρχές. Σας ευχαριστώ. The Ναι, δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι μία που δεν έχουμε ακόμα κανένα αποτέλεσμα αυτών των μελετών αντικτύπου, εμείς θα προτείναμε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά για να διατηρήσουμε τον έλεγχο και να ε, κοιτάξουμε τις εξελίξεις και να ασχοληθούμε με αυτές. Ε, να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Anybody else? Άλλος κανείς? Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ δεν συμφωνώ με τη συνάδελφο στην Ιταλία υφίστανται τόσες πολλές διαφορετικές γραφειοκρατικές νομοθεσίες για την προστασία πολλών διαφορετικών πραγμάτων και αυτή τη, στιγμή που βλέπ, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι μειώνονται όλο και περισσότερες επενδύσεις. Αυτή τη στιγμή τον επιβαρύνουμε ακόμα περισσότερο την όλη διαδικασία, η οποία από μόνη της, όπως μας είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή τη στιγμή δεν συνιστά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας και σε καμία περίπτωση δεν στρέφεται κατά της κοινοτικής οδηγίας για τους σκοτόπους. Θεωρώ λοιπόν θα ήταν πάρα πολύ ζημιογόνο εμείς αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουμε περαιτέρω γραφειοκρατικές διαδικασίες. Σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο στην Ιταλία υπάρχουν πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας, ενδεχομένως και υπερβολικές ορισμένες φορές. Νομίζω λοιπόν ότι σε εθνικό επίπεδο υφίσταται και ισχύει η εθνική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει εμείς να επιβαρύνουμε περισσότερο την όλη διαδικασία μέσω της αναφοράς αυτής και εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω λοιπόν ότι ε, αν οι ίδιες Ιταλικές αρχές κρίνουν κάποια στιγμή στο μέλλον το έργο αυτόν επικίνδυνο για το περιβάλλον, οι ίδιες μόνες τους θα αποφασίσουν τελικά ότι δεν πρέπει να υλοποιηθεί το έργο αυτό. επομένω προτείνω να κλείσει αυτή η αναφορά. Μα δείτε ότι σύμφωνα με αυτά που είπε η Κομισιόν. Η Περιφερειακή Υπηρεσία Περιβαλλοντολογικής Προστασίας απεφάνθη ότι η μελέτη που υπέβαλε ο κατασκευαστής δεν είναι αρκετά σωστή για να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς την αποτίμησή μας και λέει ότι μάλλον θα οδηγήσει σε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για το Natura 2000, για αυτόν τον τόπο του Natura 2000. Αυτό που μας είπε μόλις η Επιτροπή δηλαδή δεν έχει υπάρξει παραβίαση του ενωσιακού νόμου, αλλά θα μπορούσαμε να στείλουμε επιστολή στις αρχές λέγοντας ότι έχουμε λάβει μια αναφορά που λέει τα εξής και έτσι να την κλείσουμε. Αλλά όπως και, την προηγούμενη, και στην προηγούμενη να, του, να μάθουν ότι το παρακολουθούμε και το προσέχουμε. Μου το κάνουμε αυτό. Επιστολή, επιστολή απλή. Μπορούν να την προσέξουν αν θέλουν ή μπορούν να τη βάλουν στον κάλαθο των αχρήστων αν θέλουν. Τουλάχιστον όμως θα γνωρίζουν ότι το συζητάμε, το συζητήσαμε. Εντάξει, μάλιστα, μάλιστα. Κυρία Πρόεδρε, έχετε το λόγο, με συγχωρείτε. Συμφωνώ. Συμφωνώ ότι είναι καλό να του στείλουμε μία επιστολή. Πρωτού όμως λάβουμε την απάντησή τους, θα ήταν περίεργο εμεί να κλείσουμε αυτή την αναφορά. Δεν θα συμφωνούσα λοιπόν με τη μέθοδο αυτή να στείλουμε μια επιστολή και παράλληλα να κλείσουμε την αναφορά. Α στείλουμε την επιστολή αυτή και διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά προκειμένου να αποφασίσουμε μόνο στη συνέχεια, αφού λάβουμε δηλαδή την απάντηση και με βάση την απάντηση αν θα κλείσουμε ή όχι την αναφορά. Όχι όμως πρωτήτερα. Βλέπω ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων αυτή τη στιγμή στην αίθουσα. Σας προτείνω το ακόλουθο. Να στείλουμε μια επιστολή στις Ιταλικές Αρχές, λέγοντας τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά μέχρι να λάβουμε μια κάποια απάντηση. Αυτό σας προτείνω. Συμφωνείτε? Πολύ ωραία. Για την επόμενη αναφορά με χαρά καλωσορίζω ε, τον κύριο Φρανσίσκο Μοντόγια Τζόγια. Ε, Αναφέροντα, δεν ξέρω αν σωστά είπα το όνομά σας, καλωσορίσατε θερμά. Εκπροσωπείτε την Ένωση Κολεκτίβο ε, Ορνηθολόγικο όρνοθολογικό Σύλλογο του Μαύρου Πελαργού στην Ισπανία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Η αναφορά αυτή έχει να κάνει με ένα παλιό έργο. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Δέκα χρόνια μας απασχολεί και έχει να κάνει με την ε, ε, διασύνδεση Ισπανίας-Μαρόκου. Το 2006 είναι για ηλεκτρικό ε, έργο διασύνδεση, είναι υψηλή τάσεως από το Γιβραλτάρ, Χάιν και Μαρόκο. Είναι Natura 2000 ε, η περιοχή αυτή, το, η πλάγια Ντελοσλάτσες. Το έτος 2011 ήδη έγινε μια κοινοβουλευτική ερώτηση και ρωτούσαμε τα αντισταθμιστικά μέτρα πώς έχουν και αποκατάσταση που δεν έγινε. Ε, αντί να υπάρξουν αυτά τα μέτρα, μπορούμε να δούμε ε, ότι γίνεται ε, μια κατασκευή ε, βιολογικού καθαρισμού και κάποια άλλα έργα καταπολέμησης ε, κάποιων χωροκατακτητικών ειδών. Η Ισπανική ΔΕΗ, ο διαχειριστής του δικτύου, έπρεπε να κάνει αυτά τα έργα, το ηλεκτρικό δίκτυο της Ισπανίας, δεν το έκανε ήδη από το 2005 και προσπαθεί να το αποφύγει και να υποκαταστήσει τα αντισταθμιστικά μέτρα. Λέει ότι α, δεν μπορέσαμε να κάνουμε βιολογικό καθαρισμό, α, δεν μπορέσαμε να αγοράσουμε τα απαραίτητα χωράφια κτλ. Και έρχονται τώρα να κάνουν ένα καινούριο έργο ε, αλλά θα πρέπει να ε, μελετήσουν την κλιματική αλλαγή και το ε, διάδρομο που χρησιμοποιούν τα αποδημητικά πτηνά ε, από την Ισπανία προς το Μαρόκο. Η έκταση αυτή ονομάζεται Finca del Camoro και καλύπτει τη μισή επικράτεια της κοινότητας Ταρίφα. Ε, είπαμε λοιπόν και ζητούμε από την Επιτροπή να απαντήσει ε, στην αναφορά μας, στην ερώτησή μας, να δούμε αν τα μέτρα αυτά ε, που θα αποζημιώσουν και θα αποκαταστήσουν τη ζημία είναι νόμιμα. Και το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας απάντησε ότι βεβαίως ναι, έχουν εγκριθεί τα μέτρα αυτά και τα νέα μάλιστα που ήρθαν να αντικαταστήσουν τα παλαιότερα για το έργο αυτό. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει περιβαλλοντική μελέτη, περιβαλλοντικό αντικτύπου δηλαδή, για το έργο αυτό. Η απάντηση που μας δόθηκε είναι ναι, ότι ναι, ναι, έχει γίνει μελέτη, κανείς δεν την έχει δει, ούτε το Υπουργείο τη γνωρίζει, ούτε κανένας άλλος. Ε, πώς έχει λοιπόν η κατάσταση. Το αρχικό έργο κατέστρεψε έναν τόπο που είναι ε, ε, στη Natura 2000 και αντί να αποκαταστήσουν ε, αυτά που ήταν σημαντικά για το περιβάλλον, αποφάσισαν να κατασκευάσουν ένα νέο έργο στην ίδια προστατευόμενη περιοχή με τέλειως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τέσσερις οικότοποι ήταν στην αρχιβιότοπη μάλλον αυτοί που πλήττοντο. Με το δεύτερο έργο έχουμε άλλους τόπους ε, που πλήττονται χωρίς να ξέρουμε τι ε, δίκτυπο θα έχει όλο αυτό στο περιβάλλον και στο βιότοπο. Ε, είναι καινούργιο το έργο που κατασκευάζεται, επαναλαμβάνουμε, χωρίς μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Στο Δήμο της Ταρίφα δεν υπάρχει σχέδιο ε, πολεδομικό, χωροτακτικό ή και αν υπάρχει δεν έχει μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Και δεν ξέρουμε αυτά τα μέτρα που θα έρθουν να αποζημιώσουν τη βλάβη στο περιβάλλον αν πραγματικά είναι ε, αποτελεσματικά ή αν κάνουν χειρότερη ζημιά για τους πολίτες και για το περιβάλλον. Ο Δήμος της Ταρίφα δεν έχει ιδέα, δεν έχει ούτε μελέτη αντικτύπου, ούτε τίποτα. Δηλώνουν οι αρμόδιοι για το έργο ότι υπάρχει μια έκθεση του Δήμου, αλλά αυτή η έκθεση δεν είναι κανονική μελέτη αντικτύπου. Και ο διαχειριστής του ηλεκτρικού δικτύου στην Ισπανία ε, ανάθεσε σε ένα ίδρυμα να κάνει μια απογραφή των ειδών των πτηνών που αποδημούν και περνούν από την περιοχή εκεί. Και το χειρότερο όλων για μας ποιο είναι, ότι αυτό το δεύτερο έργο που απορρέει από το πρώτο, ας πούμε, η κατασκευή γίνεται με κοινοτικά κονδύλια. Και ο κατασκευαστής έχει αναθέσει το έργο αυτό σε μια εταιρεία, σε μια, ένα ίδρυμα το οποίο παίρνει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το θέμα αυτό δεν λύνεται σε εθνικό επίπεδο. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια πηγαίνουν σε αυτό το έργο το οποίο είναι και πάρα πολύ βραχυπρόθεσμο. Ε, ξέχασα να σας πω ότι τα εδάφη εκεί ένοικαν στο στρατό προηγουμένως και είναι πολύ μικρό το διάστημα, 15 έτη και ε, ε, ε, ξέρουμε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα λεφτά αυτά θα πάνε χαμένα γιατί υπάρχει ημερομηνία λήξη αυτή η 15 ετία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν υπάρχουν εκεί ευρωπαϊκά κονδύλια, εμείς όμως έχουμε τις αποδείξεις ότι υπάρχουν. Η επόμενη διαφάνεια είναι κάπως περίπλοκη και δυσνόητη. Δεξιά είναι αυτά ε, που ζητάει η κυβέρνηση της Ισπανίας από τον αναφερόμενο ε, να χρηματοδοτήσει και τα διπλανά είναι αυτά που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή Αντί να πληρώνει ο κατασκευαστή, πληρώνουμε όλοι εμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι φορολογούμενοι. Εδώ και 10 χρόνια ζητάμε πληροφορίε, δεν μας τις δίνουν παρά μόνο μετά από καθυστερήσει, ολιγορίες ετών ολόκληρων. Και όταν αλλάζει μια μελέτη αντικτύπου ή αλλάζει το έργο, ε, υπάρχουν κάποιες συμβατικές υποχρεώσεις. Δεν μπορείς να αλλάζεις κατά το δοκούν τα αντισταθμιστικά μέτρα ή την αποζημίωση. Δεν ξέρουμε το νέο έργο λοιπόν τι επιπτώσεις θα έχει στην περιφέρειά μας. Βλέπουμε ότι οι δηλώσεις ε, για το περιβαλλοντικό αντίκτυπο είναι απλώς ε, μια απλή διαδικαστική υπόθεση, μια διεκπεραίωση. Δηλαδή, ε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν ως αρχή. Κατασκευάζουμε κάτι, καταστρέφουμε κάτι και αντί να το αποκαταστήσουμε, συνεχίζουμε την κατασκευή ενός διαφορετικού έργου και μπορεί κάποια στιγμή να επαναρθώσουμε και τη ζημιά. Ε, ενώ θα πρέπει αντίστροφα να γίνεται αυτό. Να δούμε πρώτα τι καταστροφή θα γίνει και ο κατασκευαστής να ε, επομίζεται και το κόστος. Το 2005 Έγινε μια μελέτη πολύ καλή περιβαλλοντικού αντικτύπου ως προς τις ζώνες και τις περιοχές που θα πρέπει να προστατεύονται, αλλά σας είπα άλλαξε το έργο και δεν σέβονται ούτε την οδηγία Habitat, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει μελέτη αντικτύπου και σαν να μην έρθουν αυτά, το άκρο να ποιο είναι και τελειώνω. Όλα αυτά τα πληρώνουμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ας ακούσουμε τώρα λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Καπριάνη. Yes, thank you. So... Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, να πούμε κάποια λόγια για το αρχικό έργο το οποίο ανέφερε ο αναφέρον. Το δεύτερο κύκλωμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη ξεκινήσει μια έρευνα, μια κοινοτική πιλωτική έρευνα το 2011, μετά από την υποβολή κάποιων καταγγελιών σε σχέση με το έργο αυτό και στη συνέχεια εξέτασε όλη την τεκμηρίωση, όλα τα έγγραφα τα οποία επέβαλαν οι Ισπανικές αρχές. Τώρα, το συμπέρασμα των αλήσεων των ερευνών τότε ήταν ότι δεν υπήρξε καμία σημαντική αρνητική επίπτωση όσον αφορά τους οικοτόπους ή τα είδη τα οποία προστατεύονται στην περιοχή αυτή στην περιοχή Εστρέτσο της Ισπανίας που ανήκει στο Natura 2000. Δηλαδή το έργο αυτό δεν είχε επηρεάσει αρνητικά την ακαιρεότητα του τόπου αυτού. Συνεπώς, η πιλωτική αυτή έρευνα έκλεισε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, διότι οι Ισπανικές αρχές είχαν εγκρίνει ένα σύνολο αντισταθμιστικών μέτρων λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υπήρχε τελικά αρνητικός αντίκτυπος, σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος όσον αφορά τους οικοτόπους και τα είδη, τα αντισταθμιστικά αυτά μέτρα δεν θα έπρεπε να θεωρηθούν αντισταθμιστικά στα πλαίσια του άρθρου 6 παράγραφος 4 της οδηγίας Habitat. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό για να αποφευκτεί οποιαδήποτε παρανόηση. Αργότερα οι Ισπανικές αρχές τροποποίησαν κάποια από τα αντισταθμιστικά αυτά μέτρα και αντικατέστησαν κάποια από τα αρχικά αυτά μέτρα με κάποια νέα. Ανάμεσα στα νέα αυτά μέτρα βλέπουμε και την ανάπτυξη του κέντρου αυτού για τα αποδημητικά πτηνά και την πλανητική αλλαγή. Δημιουργεί ενό έργου που έχει να κάνει με την αποκατάσταση κάποιων στρατιωτικών κτηρίων προκειμένου να δημιουργηθεί το κέντρο αυτό για τα αποδημητικά πουλιά. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες που λάβαμε, προτού συμφωνήσουν για τα νέα αυτά μέτρα, οι Ισπανικές αρχές ζήτησαν από τον ανάδοχο να δικαιολογήσει την τροποποίηση του όλου έργου και να γίνει ενδεχομένω και μία αξιολόγηση του αντίκτυπου τόσο κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του κέντρου αυτού όσο και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του κέντρου. Στο πλαίσιο του ελέγχου λοιπόν αυτού, γιατί εμείς θεωρούμε ότι ήταν έλεγχος αυτός που έκαναν οι Ισπανικές αρχές, πάλι δεν προέκυψε κανένας αρνητικός αντίκτυπος, τουλάχιστον όσον αφορά την κατασκευή του κέντρου αυτού. Συνεπώς, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών και βάσει των εγγράφων που υπέβαλε ο αναφέρον, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που θα οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι ε, το, η δημιουργία του κέντρου αυτού για τα αποδεμητικά πτηνά και την πλανητική αλληγή θα επηρέαζε αρνητικά τον τόπο αυτό που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εντοπίσει καμία παράβαση των οδηγιών Natura και συνεπώς ε, δεν προβλέπουμε εμείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβουμε δράση κατά των Ισπανικών αρχών. Thank you very much. I open the... Ευχαριστώ πολύ. Αρχίζει η συζήτηση. Ε, οι συνάδελφοι, πρώτη η Ρώσα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Λίγο σε σχέση με τα όσα ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα τον αναφέροντα. Ναι, πρόκειται για ένα δεύτερο ε, δίκτυο διασύνδεσης ε, Ισπανίας-Μαρόκου που περνάει από τα στενά του Γιβραλτάρ και ε, είπε ο αναφερόμενος ότι μπορεί αυτό να έχει να κάνει με την οδηγία Habitat. Από το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε ζήτησε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπέθρου και Θαλάσσης να κάνουν τη μελέτη αντικτύπου και η απάντηση λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Στη συνέχεια το 2012 έγινε μια δεύτερη διαβούλευση και πάλι φάνηκε από εκεί ε, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Τουλάχιστον αυτά δηλώνουν. Ε, η Ισπανία δεσμεύεται να ιδρύσει ένα κέντρο μελέτης αποδημητικών πτηνών και ε, πάλι διαβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να έχει περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Το 2013 ήρθε η απάντηση από τις αρμόδιες αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε έκλεισε το θέμα καθυστέρησα να φτάσω και ζητώ συγγνώμη. Δεν ξέρω τι νέα στοιχεία έδωσε ο αναφερόμενος, αλλά θέλω να ακούσω τους συναδέλφους ε, αν θέλετε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά ή αν πρέπει να κλείσει. Ε, που από ό,τι φαίνεται αυτό ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να με διαφωτίσετε γιατί δεν άκουσα τι είπαν οι κύριοι. Ευχαριστώ. Συμπάγιος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στα Ισπανικά. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτά που μας λέει εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτά που λέει ο αναφέρομενος. Έχω εργαστεί ε, πολύ καιρό στην Ισπανία με περιβαλλοντική νομοθεσία και μελέτες περιβαλλοντικού αντικτύπου κτλ. και γνωρίζω ότι δεν είναι πάρα πολύ αξιόπιστες αυτές οι μελέτες πάντα. Και εξ όσων κατάλαβα, από όσα μας είπε ο αναφερόμενος, αυτό που τώρα κάνουν τι είναι. Νέο έργο κατασκευάζουν εκεί, χωρίς να υπάρξει προηγούμενη μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Ε, ανεξαρτήτως ε, από τα όσα είπατε για το προηγούμενο έργο. Και τα αντισταθμιστικά μέτρα βεβαίως δεν τηρούνται. Αυτό είναι κανόνας ουσιαστικά στην Ισπανία. Ε, και τώρα εφευρίσκουν ένα νέο έργο και πάλι δεν έχω καταλάβει πολύ καλά Ποιο χρηματοδοτεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν χρηματοδοτούμε εμεί. Αλλά ε, στα πανό που έχουν βάλει εκεί και τα έχουμε δει, έχει τη σημαία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παντού. Και η ερώτηση είναι, πηγαίνουν και ευρωπαϊκά κονδύλια ή απλώς το έχουν βάλει για διαφήμιση και δεν έχει κανένα έλεγχο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Mm. Νομίζω κάποιο λάκκο έχει φάβο εδώ. Και επίσης αυτό που λείπει από τις μελέτες περιβαλλοντικού αντικτύπου στην Ισπανία είναι η εναλλακτική κατασκευή σε, άλλο, σε άλλη τοποθεσία. Δεν ξέρω εάν το έχουν ψάξει, αν μπορεί να γίνει πουθενά αλλού αυτό το έργο με λιγότερη ζημιά. Δεν το ξέρουμε, δεν υπάρχει εναλλακτική μελέτη, τουλάχιστον αυτό διαβάζουμε. Και επίσης ο αναφερόμενος ζήτησε και για, ε, μίλησε και για διαφθορά και για άσκηση πίεσης και εκφοβισμό. Γίνεται αυτό πολλές φορές στην Ισπανία. Οπότε, εγώ μάλλον θα άφηνα ανοιχτή αυτή την αναφορά. Δεν θέλω να θαυτεί. Να συνεχίσουμε να ψάχνουμε αυτό, το πώς έγινε η μελέτη αντικτύπου για ε, το έργο αυτό. Αν έχουν μελετήσει εναλλακτικέ και από πού έρχονται τα λεφτά και πού πηγαίνουν. Και θέλω να ρωτήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν έχει μεταβεί επιτόπου να κάνει έλεγχο. Εκεί, στην Ταρίφα, εκεί που θα γίνει αυτό το έργο, στην Ανταλουσία. Ή απλώ ακούτε αυτά που σας λένε οι Ισπανικές αρχές, γιατί εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Άλλο να διαβάζεις αυτά που σου στέλνουν οι κρατικές αρχές και αυτά που σου λένε και άλλο να πας να το δεις με τα ίδια σου τα μάτια. Οπότε Θέλω και εγώ να ρωτήσω αν μετέβει εκεί στην ταρήφα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαπιστώσει ισόμες στην κατάσταση. Ευχαριστώ. Κύριε Τερικα Μπράς, ευχαριστώ. Εγώ πιστεύω ότι έχει πέσει σε σημαντικές ε, αντιφάσεις ε, η κυβέρνηση ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το τις κατέριψε. Λένε ότι υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικό αντικτύπου, είπε ο αναφέρομενος, ε, ε, αλλά αυτή δεν υπάρχει. Και υπάρχουν και ευρωπαϊκά κονδύλια δεν υπάρχουν για χρήση και κατάχρηση κατά το δοκούν. Και πάλι δεν απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικές αντιφάσεις από πλευρά των Ισπανικών αρχών. Είπε η Κομισιόν ότι δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό. Αυτό το απάντησε όμως το 2011. Ενώ μας λέει ο κύριος εδώ ότι το 2012 άλλαξε η πρόταση, άλλαξε το έργο που φαίνεται ότι είναι χειρότερο από το προηγούμενο και επίση είναι περίεργο, έτσι, λίγο μυστήριο, να υπάρχουν αντισταθμιστικά μέτρα γιατί αν όλα γίνονται ωραία και καλά, τι να αντισταθμίσουν άμα δεν υπάρχει ζημιά, τι να επανορθώσουν. Για να έχεις αντισταθμιστικά μέτρα σημαίνει ότι κάποια βλάβη κάνεις εκεί, αλλιώς για ποιο λόγο. Οπότε και ειλικρινά, μέχρι να λυθούν αυτά τα πράγματα που είναι τελείως ουσιαστικά για μένα, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να κλείσει αυτή η αναφορά. Ευχαριστώ πολύ. Mr. Ο κύριος Μάτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να πάρω το λόγο γιατί νόμιζα ότι είχαν ξεκαθαριστεί μετά την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα πράγματα. Αλλά α, ακούγοντας αυτά που ακούμε εδώ μέσα νομίζω ότι καλό θα ήταν να πούμε τα εξή τουλάχιστον. Ποιο λάκκο να έχει φάβα και ποια φάβα. Δεν βλέπω εγώ τίποτα μυστήριο εδώ. Και τα λέμε έτσι πολύ ελαφρά την καρδία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στην Επιτροπή μας ότι υπάρχει εδώ διαφθορά και άσκηση πιέσεων. Δεν το λέω για την Πρόεδρο. Ε, αν υπάρχει αυτό να πάτε στον Ισαγγελέα και στα δικαστήρια. Δεν μπορούμε να λέμε στον αέρα όπως είπε μια συνάδελφος ε, συγκαλυμμένες κατηγορίες αν δεν πούμε επόμενα. Αυτό είναι αδίκημα. Εάν γνωρίζετε ότι έχει παρανομήσει κάποιος και η άσκηση πιέσεων και η ε, διαφθορά, να πάτε να τα πείτε στα δικαστήρια, αλλιώ να μην λέτε τίποτα, να σιωπήσετε. Και όταν γίνεται λόγος για εναλλακτικέ τοποθεσίες που να υπάρξει μικρότερη ζημιά, εμείς κοιτάμε εάν τηρείται ο νόμος ή αν δεν τηρείται και αντίστοιχε οδηγίες. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι απολύτως τηρείται ο νόμος. Εδώ πολλές φορές θέλουμε να ε, κάνουμε μαθήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τις αλλάξουμε ε, τη δουλειά. Εάν δεν έχει τίποτα, πώς να το πω, αν έχουν μείνει σκιές, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχει τίποτα παράνομο όταν κάποιος ε, λαμβάνει αποζημίωση είναι όταν το απατριώνουν ας πούμε ε, τη γη του για να φτιάξουν ένα έργο, μια φυλακή, ένα νεκροταφείο ή κάτι άλλο πρέπει να αποζημιωθεί ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου. Δεν υπάρχουν εδώ παρανομίες. Κάπως έχει ανάψει η συζήτηση λέει η Πρόεδρος. Έχει ανάψει η συζήτηση. Μισό λεπτό δεν σας έδωσα το λόγο. Δεν σας έχω δώσει το λόγο. Επόμενος ομιλητής. Επόμενη είναι η κυρία Αλμπιόλ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα απλώς να πω ότι εμείς θεωρούμε, ακούγοντας και το συντάκτη της αναφοράς και την κυρία Σεπάιο και τους υπολείπους, συμφωνούμε ότι υπάρχουν απολύτως επαρκή στοιχεία για να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, ιδιαίτερα γιατί η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δόθηκε το 2011, ενώ η αλλαγή του έργου έγινε το 2012 και το θέμα είναι αν έχουν χρησιμοποιηθεί ευρωπαϊκά κονδύλια ή όχι. Και μόνο αυτά τα δύο αρκούν για να παραμείνει ανοιχτή αναφορά και τουλάχιστον να διερευνηθεί αυτό το θέμα. Αυτά τα δύο ερωτήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα έχετε το λόγο. Κύριε Ταρίκα Βράς, παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη. Ήθελα απλώ να ξεκαθαρίσω ότι ε, συνέδεσε με το όνομα μου πράγματα εγώ που, ε, που εγώ δεν είπα. Εγώ δεν μίλησα για απάτη, ούτε για δικήματα ούτε για εγκλήματα, ούτε τίποτα. Θα πρέπει να κάνουμε μια καθαρή συζήτηση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Anybody else? That... Ευχαριστώ πολύ. Κανένας άλλος. Η Ρώσα. Η τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και αν να με διορθώσει, η Κομισιόν είναι 24 Ιανουαρίου 2013, είναι μετά το 12 δηλαδή. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντησή της λέγει ότι μπορεί να κλείσει αναφορά διότι όλα είναι σύνομα και σε καμία περίπτωση τα αντισταθμιστικά μέτρα δεν παραβιάζουν την οδηγία Habitat. Και 21 Δεκεμβρίου 2012 υπάρχει άλλη απάντηση που είναι μετά τα γεγονότα. Δεν ξέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπερασπιστεί τον εαυτό της, δεν χρειάζεται να το κάνω εγώ. Can give the floor for a very short comment from the... δώσω το λόγο για πολύ λίγο χρόνο μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά τώρα το νέο έργο, άκουσα ότι δεν έγινε η απαραίτητη, η κατάλληλη αξιολόγηση. Η οδηγία Habitat, αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου, δεν λέει ότι οποιοδήποτε έργο στα πλαίσια του Natura 2000 θα πρέπει να υπόκειται σε αξιολόγηση. Μόνο τα έργα εκείνα τα οποία ενδεχομένω μπορούν να έχουν σημαντικέ αρνητικέ επιπτώσει. Εναπόκειται λοιπόν στι αρμόδιε εθνικέ αρχέ να αποφασίσουν αν ένα συγκεκριμένο σχέδιο, αν ένα συγκεκριμένο έργο μπορεί πραγματικά να έχει αρνητικές επιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή ζητούν από τον ανάδοχο περισσότερες πληροφορίε, αυτό κάνανε και για τον ανάδοχο του κέντρου αυτού για τα αποδημητικά πτηνά και βάσει των πληροφοριών που στέλνει ο ανάδοχος αυτός όσον αφορά την αποκατάσταση των υφιστάμενων στρατικών κτηρίων, με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν για τον οικότοπο αλλά και για τα προστατευόμενα πτηνά, μπορούν και αποφάσισαν προκειμένου ότι δεν χρειαζόταν να γίνει μια πλήρης περιβαλλοντική αξιολόγηση. Αυτό προβλέπεται και επιτρέπεται ως ενδεχόμενο από την οδηγία Habitat. Τώρα, αν να αναφέρον θέλει να καταγγείλει μια τέτοια πρακτική θα πρέπει να προσκομίσει και αποδεικτικά στοιχεία. Τέτοια αποδεικτικά στοιχεία δεν φτάσαν σε εμά που να δείχνουν ότι πραγματικά μπορεί να υπάρχει πραγματικό αρνητικό αντίκτυπο στο συγκεκριμένο οικότοπο ή στα πτηνά τα οποία ζουν στην περιοχή αυτή. Συνεπώ εμεί δεν μπορούμε να γύρουμε τέτοιο ζήτημα με τι πανικέ αρχέ. Δεν πήγαμε προφανώ γιατί δεν ήταν αναγκαίο πρώτον και δεύτερον γιατί δεν κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε εμεί αρμοδιότητε επιθεώρησης. Εμείς μπορούμε να γύρουμε το ζήτημα αυτό μόνο αν λάβουμε αποτεκτικά στοιχεία από οποιαδήποτε πηγή. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, να δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου από την DG Agri. Γεια σας, Ερνάντες λέγομαι, πολύ σύντομα. προσωπώ τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και ε, Ανάπτυξη Υπέθρου. Χωσέ Μανουέλ Ερνάντε. Για τη χρηματοδότηση, πολύ γρήγορα. Είχαμε πρόσβαση βεβαίως στη χρηματοδότηση πολύ σύντομα, πριν από λίγες μέρες, πολύ πρόσφατα μάλλον, και φαίνεται ξεκάθαρα ε, ότι συμμετέχει το ΦΕΝΤΕΡ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μέχρι τώρα δεν έχουμε συγκεκριμένα ε, στοιχεία ότι χρηματοδοτήθηκε από κοινοτικά κονδύλια, αλλά εφόσον υπάρχει και αυτό το πανό, προφανώς έχει χρηματοδοτηθεί από κοινοτικά κονδύλια. Και το ΦΕΝΤΕΡ χρηματοδοτεί κάποια έργα τα οποία χειρίζονται τα κράτη-μέλη. Εκείνοι κάνουν τους ελέγχους, εκείνοι εκτελούν τον προϋπολογισμό και όπως είπε και ο συνάδελφος από το περιβάλλον, κάθε έργο το οποίο ενδεχομένως να επηρεάζει σημαντικά το περιβάλλον θα πρέπει να υπόκειται σε μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Και αυτά τα χειρίζονται ε, οι αρμόδιες αρχές της κάθε χώρας, του κάθε κράτους μέλους. Αυτοί κάνουν και τον έλεγχο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ενέχεται στην επιλογή ούτε στον έλεγχο των όρων. Εδώ ισχύει επικουρικότητα. Το πολύ πολύ που μπορεί να κάνει οικονομικό έλεγχο για να δει αν έχουν κατάλληλα συστήματα ελέγχου και κατάλληλα μέτρα για το λογιστικό έλεγχο, επαναλαμβάνω, τα κράτη-μέλη. Μόνο μετά από κοινοβουλευτικέ ερωτήσεις ή από αναφορές μπορούμε εμείς να επέμβουμε ή να απαντήσουμε. Προφανώς καθημερινά δεν μπορούμε να παρακολουθούμε την επιλογή, την ε, κατασκευή, την πορεία κάθε έργου. Αυτό μόνο ήθελα να διευκρινίσω. We are actually running έχουμε καθυστερήσει. Μήπως υπάρχει κανείς άλλος που θέλει να κάνουμε τίποτα άλλο. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχουμε διαφορετικές απόψεις για το θέμα, άρα δεν μπορώ να το κλείσω. Δεν γίνεται. Αφού οι διάφοροι ομιλητές είπαν ότι θέλουν να παραμείνει η αναφορά ανοιχτή. Και άρα η γραμματεία πρέπει να προσπαθήσει να βρει έναν σωστό τρόπο προώθησης. Γιατί να μείνει απλώς ανοιχτή δεν είναι λύση, εκτός αν ξέρουμε τι άλλο χρειάζεται. Θα τη δώσουμε λοιπόν στη γραμματεία για να ερευνήσει περαιτέρω εάν χρειάζεται να κάνουμε τίποτε άλλο. Θα ήθελα εξάλλου να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την πληρέστατη απάντησή της. Τα κοίταξε όλα με λεπτομέρεια φαίνεται. Και παρόλα αυτά οι συνάδελφοι, μερικοί συνάδελφοι θέλουν και άλλες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πάντως για όλες εκείνες τις πληροφορίες που μας δώσατε και τώρα η γραμματεία μας θα προσπαθήσει να βρει τι άλλο βήμα πρέπει να γίνει. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον αναφερόμενο για να σχολιάσει εκεί στο τέλος. Με μικρόφωνο παρακαλούμε. Όπως σας είπα προηγουμένως και ακούστηκε και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κανονικά, ε, ο, ο ανάδοχος ε, έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Εκείνος προτείνει τα αντισταθμιστικά μέτρα, εκείνος προτείνει τις μελέτες. Αλλά εμείς δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο ανάδοχος έχει τον πλήρη έλεγχο των κινήσεων. Αλλά δεν μπορεί να, να βγει και να αυτοκατηγορηθεί και να πει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον το έργο του. Είναι κριτής και κρινόμενος. Μάλιστα. Η γραμματεία θα ε, συνεχίσει να ε, μελετάει και να ερευνά το θέμα αυτό. Ευχαριστώ που ήρθατε να μοιραστείτε μαζί μας ε, τις απόψεις σας και τις εμπειρίες. Δεν κλείνει η αναφορά, διατηρείται ανοιχτή και θα επανέλθουμε εν ευθέτω χρόνο. Επόμενη αναφορά. Σχετικά με τα λύματα στην περιοχή Μονκόφα της Ισπανίας. Πολλά ισπανικά θέματα έχουμε υπερβαλλοντικά. Είναι υπαριθμόν 1260 σημείο 8. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε τον κύριο Φερνάντες Γκόμες και με πολύ χαρά σας δώσω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Στην αναφορά αυτή περί τίνος πρόκειται. Δεν υπάρχει επεξεργασία λιμάτων. Λατόρε λέγεται ε, ο οικισμός και υπάρχει και ένα κάμπινγκ εκεί. Παράγουν λίματα που δεν υφίστανται επεξεργασία. Αυτά ε, τα νερά πηγαίνουν ε, σε μια λεκάνη καθίζησης και μετά μεταφέρονται υποτίθεται σε μια έκταση που έπρεπε να ε, είναι ε, η επεξεργασία, βιολογικός καθαρισμός. Λιμνάζουν όμως και πηγαίνουν σε ένα κανάλι, ε, υποδηγεί σε φράγμα και μετά στη θάλασσα αυτά τα βρώμικα λίματα θεωρεί ο αναφερόμενος ότι μπορεί να επηρεάσουν ε, τα ύδατα κολύμβηση σε μια κοντινή παραλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελέτησε ε, όλες αυτές τις πληροφορίες και από ό,τι φαίνεται ότι ε, ο οικισμός αυτός είναι μικρός ή πάση περιπτώσει είναι λιγότερο από 10.000 οι κάτοικοι και βάσει του άρθρου 7 της Οδηγίας 91-271 Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα λίματα. Όταν πρόκειται για οικισμούς που έχουν λιγότερους από 10.000 κατοίκους θα πρέπει να υφίστανται ένα ε, είδος επεξεργασίας ε, ανάλογα με την κοινοτική νομοθεσία και μάλιστα όλα αυτά έπρεπε να γίνουν μέχρι το τέλος του 2005. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης διαπίστωσε ότι για το 2013 η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην ε, παραλία ε, ε, θεωρείται εξαιρετική, ιδιαίτερα ήδη από το 2008. Φαίνεται επομένως ότι δεν επηρεάζεται από τις απορρίψεις ε, των λιμάτων αυτών η ποιότητα των υδάτων κολύβησης. Η Επιτροπή λαμβάνει γνώση της κατάστασης. Αυτό τον καιρό κατασκευάζεται μια μονάδα ε, βιολογικού καθαρισμού στην πόλη Μονκόφα που τους επόμενους μήνες θα τεθεί σε λειτουργία. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία, δηλαδή το μικρό μέγεθος του οικισμού, το μικρό αριθμό των κατοίκων, ε, τα περιορισμένα λίμματα και το γεγονός ότι δεν επηρεάζουν τα ύδατα κολύμβησης αλλά και ότι έχει δρομολογηθεί λύση, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην παρέμβει για το θέμα αυτό Είναι προτεραιότητα η επεξεργασία των λιμάτων και τώρα αυτό το καιρό υπάρχουν διάφορες διαδικασίες που τρέχουν. Υπάρχει και καταδίκη της Ισπανίας από το 10 για μη σωστή εφαρμογή της οδηγίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε λοιπόν να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στις διαδικασίες αυτές που έχουν δρομολογηθεί, να προχωρήσουν δηλαδή και αντί να δούμε μεμονωμένα αυτή την περίπτωση, γιατί είναι και ίσονο σημασία, μάλλον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Thank you. And the floor is open for... Ευχαριστούμε. Μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση. Ο Αλμπιόλ Γκούσμαν. Παρακαλώ. Eh, Ευχαριστώ. Οι αναφερόμενοι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν. Ζήτησα να μπορέσω εγώ να τους εκπροσωπήσω. Πράγμα που θα κάνω γιατί τους έχω συναντήσει ε, αυτή την Ένωση των Κατοίκων πριν από λίγους μήνες. Ξέρω το πρόβλημα, ξέρω και την κατάσταση και εγώ από εκεί κατάγομαι, από την επαρχία Καστεγιών στην Ισπανία και θέλω να υπερασπιστώ αυτή την υπόθεση. Περί τίνος πρόκειται. Είναι 2.000 τα σπίτια εκεί, αλλά υπάρχει και κάμπινγκ και μια βιομηχανική ζώνη. Οπότε δεν είναι μόνο τα 2.000 σπίτια, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι περισσότεροι οι ε, άνθρωποι και τα ζητήματα. Ε, τα ε, λίματα πηγαίνουν κατευθείαν στη θάλασσα, γιατί δεν είναι μονάδα βιολογικού καθαρισμού, είναι απλώς μια μονάδα καθίζησης η οποία καταραίει, γιατί κατακλείζεται από τα βρώμικα νερά αυτά και πηγαίνουν και σε ένα κανάλι υδάτων. Και όταν ξεχυλήσει βγαίνουν λοιπόν τα λίμματα ε, σε κανάλι ομβρίων υδάτων και καταλήγουν στη θάλασσα. Είναι υπόνομος ουσιαστικά. Και αυτό τι σημαίνει. Υπάρχει κίνδυνος και για τη δημόσια υγεία και επίσης έχουν ας πούμε τα παιδάκια ε, δερματικά προβλήματα όταν κάνουν μπάνιο στη θάλασσα και το αποδίδουν ε, άμεσα σε αυτό οι κάτοικοι. Και επίσης ε, υπάρχουν βλάβες και για το περιβάλλον αλλά και γενικότερα προβλήματα για τον τουρισμό. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για τουριστική περιοχή, παραθαλάσσια και έχει και γαλάζια σημαία η παραλία πολύ κοντά που έχει δοθεί από τον αρμόδιο ευρωπαϊκό φορέα και μπορεί να πληγεί και η εικόνα και ε, γενικότερα το όνομα της περιοχής. Υπάρχουν διάφορες οδηγίες, μια οδηγία για τα λίματα, τα αστικά, υπάρχει μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα λίματα επίσης και για την γενικότερη οδηγία ε, των υδάτων. Υπάρχουν λοιπόν αρκετοί λόγοι έτσι ώστε να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι κάνει. Νύπτει τα τη. της. Ε, σου λέει είναι πάρα πολύ μικρό ο οικισμός για να ασχοληθώ. Αλλά το καλοκαίρι πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμό. Δεν είναι ε, όσοι έχουν συμπεριληφθεί στην απογραφή. Και 5.000 μπορεί να βρει κανείς εκεί. Και επαναλαμβάνω υπάρχει και κάμπινγκ εκτός από τον οικισμό εκεί και ε, τρία μεγάλα εργοστάσια ε, κεραμικής που χρησιμοποιούν πάρα πολύ νερό και βεβαίως χωρίς καθαρισμό ε, ρίχνουν τα λίματα μαζί με τα υπόλοιπα του υπονόμου. Το ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαλείται το βιολογικό καθαρισμό. Δεν υπάρχει καθαρισμός, είναι ένας βόθρος που καταλήγει στη θάλασσα ουσιαστικά σε τουριστική περίοδο, σε τουριστική περιοχή. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει για τα ξενοδοχεία και για τον τουρισμό. Μας λένε ότι κατασκευάζεται βιολογικός καθαρισμός χρόνια τώρα, έχει οδηγηθεί σε παράλυση, έχει αποτελματωθεί ουσιαστικά, ούτε προβλέπετε πότε θα ολοκληρωθεί, γιατί τους έχουν τελειώσει τα λεφτά ε, στο Δήμο και ξέρετε τι γίνεται ε, με τα δημόσια ταμεία στην Ισπανία και την κοινότητα, ε, την αυτόνομη περιφέρεια της Βαλένθια, δεν έχει λεφτά ε, για να ολοκληρώσει το έργο και για να λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός. Η μονάδα επεξεργασίας λιμάτων. Το έχουμε πει αυτό και στο Μογκόφαρ και στην περιφερειακή κυβέρνηση της Βαλένθια. Θα πρέπει να στείλουμε κι εμείς ως Επιτροπή μία επιστολή για να ρωτούμε τι γίνεται και προς το Δήμο και προς την κυβέρνηση της Βαλένθια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακούσαμε τη συμπροματική προφόρηση της ε, κυρίας Αλμπιόλ. Εάν προβλέπεται να ολοκληρωθεί η μονάδα επεξεργασίας λιμάτων, δεν μπορούμε να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο και να αρχίσει να λειτουργεί. Του, τουλάχιστον. Και ακριβώς αφήνοντας ανοιχτή την αναφορά μπορεί και να επιταχυνθεί η εκτέλεση του έργου, πράγμα που είναι ευχής έργων για το περιβάλλον. Εγώ θα προτιμούσα να περιμένουμε και να δούμε τι θα γίνει με τη μονάδα επεξεργασία που μπορεί να έχει πολύ μεγάλη σημασία για μια τέτοια περίπλοκη περίπτωση. Ναι, εγώ διαφωνώ. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ενημέρωσε σαφέστατα και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα ύδατα κολύμβησης. Ε, η κυβέρνηση της Ισπανίας είπε ότι προσεχώς θα αρχίσει να λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός και εμείς εδώ είμαστε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είμαστε Περιφερειακό Κοινοβούλιο στην αυτόνομη περιφέρεια. Να το θέσει εκεί η κυρία Αρμπιόλα, έχουν και πολλές αρμοδιότητες οι τοπικές βουλές στην Ισπανία. Η ευρωπαϊκή αρμοδιότητα είναι σαφέστατη και είπε η Κομισιόν ότι είναι εντάξει, δεν παραβιάζεται κοινοτική οδηγία και δεν θίγονται τα ύδατα. Τώρα θα περιμένουμε εμεί να γίνει ο βιολογικό καθαρισμό. Αυτό είναι τοπική αρμοδιότητα τη περιφέρεια, δεν τη Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι από ευρωπαϊκής πλευράς είμαστε εντάξει. Εγώ θα έλεγα να κλείσει αναφορά, πράγμα που δεν σημαίνει ότι απαγορεύει κάποιο να γίνει συζήτηση σε περιφερειακό επίπεδο, που σε αυτό αναλογεί όμω, όχι σε ευρωπαϊκό. Έχουν εκχωρηθεί οι ε, αρμοδιότητες στην περιφέρεια και σε αντίθετη περίπτωση είναι σε εθνικό επίπεδο, αλλά όχι σε ευρωπαϊκό. Θα πρέπει να κλείσει λοιπόν η οδηγία ευχαριστώ. Μετά την ενημέρωση της κυρίας Αλμπιόρ έχει σημασία να δούμε τι είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μιλάει για τις μελέτες που έγιναν στα είδατα κολύμβησης το 2013. Για το 2014 έχετε στοιχεία γιατί ένας χρόνος είναι αρκετό διάστημα και μεγάλο μάλιστα και σίγουρα θα έχει υπάρξει αλλαγή και μπορεί αυτή η πληροφόρηση να μας βοηθήσει για να υπάρξει δράση σε επίπεδο Δήμου και σε επίπεδο περιφέρειας. Ε, αλλά το ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και αν κλείσει αναφορά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μελετήσει την ποιότητα των υδάτων και για το 14, όχι το 2013. Μισά Η κυρία Αλμπιόλ. Ναι, ευχαριστώ. Συμφωνώ. Τουλάχιστον να μείνει ανοιχτή η αναφορά μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο το ξέρω ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά ένα από τα επιχειρήματα της Επιτροπής είναι ότι σε λίγο καιρό θα αρχίσει να λειτουργεί η μονάδα επεξεργασίας λιμάτων. Ναι, αν είναι αυτό ένα επιχείρημα για να κλείσει ένα φορά είναι εξίσου επιχείρημα για να διατηρηθεί ανοιχτή, γιατί λέμε ότι δεν έχει κατασκευαστεί ακόμα. Και χρειάζεται τα λύματα να έχουν τον κατάλληλο βιολογικό καθαρισμό. Μα δεν είναι κατάλληλο καθαρισμός να πηγαίνουν να χύνονται στη θάλασσα αυτά τα βοθρολήματα όπως βγαίνουν. Το είπε και η κυρία Πεσέρα, να δούμε τι γίνεται με το 14 και να περιμένουμε να ολοκληρωθεί το έργο και μετά να κλείσει αναφορά. Mr. Ο κύριος Τάρη Ευχαριστώ. Με κάλυψε η, κυρία Αλμπιόλ. Αυτό το επιχείρημα είχα να πω και εγώ για τη μονάδα επεξεργασίας. Κύριε Σεμπαστιά. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Είναι ένα θέμα που το ήξερα και έχω τη δυνατότητα και εγώ να το επιβεβαιώσω. Βεβαίως και είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ποιότητα των υδάτων και επαγρύπνηση και για να γίνει αυτό, ο μόνος τρόπος που υπάρχει είναι να συμμορφωθούν και για να συμμορφωθούν πρέπει να κατασκευαστεί αυτή η μονάδα βιολογικού καθαρισμού. Δεν μπορεί να κλείσει η αναφορά. Έχουν ευθύνη τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Πρώτον, χρειάζεται μια μελέτη πιο πρόσφατη για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης και αν η δικαιολογία για να κλείσει η αναφορά είναι ότι ο Σονούπο θα αρχίσει να λειτουργεί η μονάδα, ε, πότε υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία μόνο όταν το ξέρουμε αυτό, τότε θα την κλείσουμε και όχι νωρίτερα. Δεν βλέπω άλλους ομιλητές. Υπάρχει κάποιος που θέλει το λόγο, παρακαλώ. Όπως και με την προηγούμενη αναφορά, Έχω την εντύπωση ότι είμαστε στην Ισπανία σήμερα. Όλοι μιλάνε Ισπανικά. Γινόμαστε μια Ισπανική επιτροπή. Ωραία λέγει αυτή. Μακάρι τα πράγματα να ήταν τόσο καλά, ή μάλλον ο καιρό να τόσο ωραίο όσο στην Ισπανία, όταν θα τελειώσουμε τη συνεδρίασή μα. Λοιπόν, τι κάνουμε με την αναφορά αυτή. Οι συνάδελφοι έχουν ζητήσει να διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά και θα ζητήσουμε μία επικαιροποιημένη ανάλυση της κατάστασης και θα ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις, τα τελευταία στοιχεία για την ποιότητα του νερού. Και επίσης θα ζητήσουμε από τις πανικές αρχές να μας πούνε τι προτίθεται να κάνουν προκειμένου να διασφαλίσουν ασφαλές νερό για τους πολίτες. Ξέρετε ότι Μπορεί να υπάρχει αυθονία νερού, μπορεί το νερό να είναι περιορισμένης ποσότητας, πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό να υφίσταται ασφαλές νερό, να παρέχεται ασφαλές νερό για τους πολίτες. Συμφωνείτε λοιπόν με αυτή την προσέγγιση. Πολύ ωραία. Περνάμε στην επόμενη αναφορά, η οποία άκουσον άκουσον είναι και αυτή η ισπανική. Και έχει να κάνει με την καταστροφική για το περιβάλλον διαχείριση της λεκάνης του ποταμού Τάγου. κυρία Βαλίνας είχε υποβάλει το αίτημα αυτό, επομένως δίνω κατευθείαν το λόγο σε εσά. Έχουμε όμως και τους αναφέροντες μαζί μας. Καλωσορίσατε, σε ζητώ συγγνώμη. Δεν κοιτούσα το σωστό εγγραφό. Κυρία Ρώσα Πριετρούης και ο κύριος Μιγγέλ Άγχελ Σάνσες Περές είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Σας ακούμε λοιπόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που μας καλέσατε στην Επιτροπή σας για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε πώς έχει η κατάσταση που είναι πραγματικά οριακή του ποταμού Τάγου. Επίσης, αισθανόμαστε απροστάτευτοι όσοι ζούμε στις όχθες του ποταμού αυτού. Ο Ντανιέλ Μαρτίνεθ είναι ο περιφερειακός ε, συντονιστής της Ενωμένης Αριστεράς και μαζί από το 2012 κάναμε αυτή την αναφορά. Ε, είχαμε χάσει όλες τις ημερομηνίε. το 2014 επανήρθαμε γιατί το σχέδιο ε, αυτό που θέλανε να υλοποιήσουν δεν είχε λάβει υπόψη τους σηκωτόπους. Επανερχόμαστε σήμερα γιατί το Σεπτέμβριο του 2014 η Ισπανική κυβέρνηση εξέδωσε ένα βασιλικό διάταγμα ε, ερήμην των πολιτών είχε συμφωνηθεί χωρίς προηγούμενη δημόσια διαβούλευση και ε, αφήνει το ποτάμι εκτός του σχεδίου του υδραλογικού για την Κουέγκα. Ο τάχος ποταμός λοιπόν ε, λέει ότι δεν πρόκειται να δέχεται πάνω από 365 ε, κυβικά εκατόμετρα το χρόνο. Το 80% του καθαρού νερού πηγαίνει σε ιδιωτικά συμφέροντα στην Ανατολική Ισπανία σε σχέση με τη λεκάνη απορροής. Γιατί ερχόμαστε εδώ. Γιατί το κανάλι που μεταφέρει ε, από τον τάγο και εκτρέπει 12 ε, κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο, ενώ στο Αραχουέθ, την πόλη αυτή, το ε, ποτάμι κατεβάζει 6 κυβικά το δευτερόλεπτο. Ο κύριος Άριας Κανιέτε έχει κάνει ένα σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής, αλλά προσπαθεί να παρακάψει ε, την οδηγία πλαίσιο για τα πτηνά. Και έχουμε έρθει σήμερα γιατί ο δεύτερος κύκλος προγραμματισμού που μόλις άρχισε στο κράτος της Ισπανίας όχι απλώς ε, διατηρεί τα δεινά του προηγούμενου σχεδίου αλλά έρχεται να τα επιδεινώσει έτσι περαιτέρω μόνο το 20% των υδάτων ελέγχονται από την εκτροπή ε, του τάγου. Σήμερα ερχόμαστε γιατί καθυστερούν ακόμα περισσότερο τις ημερομηνίε ε, στις οποίες θα πρέπει να καταθέσουν τις μελέτες για την καλή κατάσταση των υδάτων. Λοιπόν, η κατάσταση του ποταμού είναι πραγματικά ωριακή. Βλέπετε ε, τη διαφάνεια. δεν φτάνει το νερό. Ή το νερό θα πάει στην Ανατολική Ισπανία ή θα μείνει στο ποτάμι, αλλιώ θα στερέψει. Είναι κατάφορο ε, παράδειγμα στην Ευρώπη ολόκληρη για παραβίαση της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχει έρθει η ώρα για την πολιτική της δράσης. Έχει έρθει η ώρα να αποφασίσει κανείς εάν πραγματικά είναι με το περιβάλλον ή με τα οικονομικά συμφέροντα και ε, τα ιδιωτικά συμφέροντα της Ανατολικής Ισπανίας. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποδείξει ότι ενδιαφέρει η οδηγία για τους οικοτόπους, για τα πτηνά και για τα ύδατα. Για να δούμε αν θα την επιβάλλουμε αυτή. Οι Ισπανοί και Πορτογάλοι ε, πολίτες που ζουν στις όχθες του ποταμού Τάγου ερχόμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε το νερό του ίδιου μας του ποταμού, που θέλουμε να παραμείνει ζωντανό το ποτάμι μας και να μην στερέψει. Ευχαριστώ πολύ και δίνω αμέσω το λόγο στο συνάδελφο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που ερχόμαστε και σας πιέζουμε σήμερα τόσοι Ισπανοί, αλλά και εσείς θα πρέπει να αναρωτηθείτε γιατί έχουμε έρθει τόσοι πολλοί Ισπανοί και ζητάμε τη βοήθειά σας εδώ. Δεν θέλουμε να στερέψει αυτό το ποτάμι. Βλέπετε τις φωτογραφίες που σας δείχνουμε. Είναι η πόλη του Τολέδο, παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και Αρανχουές επίσης, ε, σπουδαία πόλη. Το ποτάμι αυτό έχει πεθάνει, έχει στερέψει, ε, μαζεύει λίματα και όπως είπε η συνάδελφος, ε, από την κήτη του ποταμού και από την πηγή του είναι σημαντικό σόγκος νερού έχει εκτραπεί που κατά την άποψή μας δεν συνάδει αυτό με κάποιες ευρωπαϊκές οδηγίες. Είναι οδηγία για τα ύδατα, για τα πτηνά, για τον οικότοπο. Και ούτε για την Ισπανική κυβέρνηση, γιατί η Ισπανική κυβέρνηση έχει δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014 ένα σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης και έχει προχωρήσει και σε τροποποίηση της νομοθεσίας. Και πραγματικά βγάλανε ένα βασιλικό διάταγμα για να παρακάμψουν όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή δηλώνουν κάτι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ισπανία κάνουν κάτι διαφορετικό για να γίνει το ποτάμι σε αυτή την κατάσταση που βλέπετε. Και επίσης αυτή την αναφορά ως ε, αναφερόμενη την έχουμε υποβάλει από το 2013 με τα αντίστοιχα στοιχεία Και μαζί με τη σημερινή ερχόμαστε να ε, σας πούμε ότι περιμένουμε απάντηση. Η Ισπανική κυβέρνηση ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει. Δηλαδή, κοιτάξτε αυτή τη φωτογραφία. Πάνω είναι λίματα από τη Μαδρίτη. Και έχουν κάνει το τάγο αυτό το ριάκι που βλέπετε κάτω. Και σας δηλώνει και ότι έχει σχέδιο γιατί κάνει λεκάνη απορροής. Το ποτάμι μας πεθαίνει και γεμίζει λίματα. Φυσικά δεν μπορούμε να πάρουμε νερό πόσιμο γιατί δεν πίνεται το νερό, ούτε για άρδευση γιατί δεν έχει νερό και όταν έχει νελίματα και ακόμα λιγότερο για κολύμβηση. Καμία περίπτωση. Η Ισπανική κυβέρνηση, το, σημερινό Λαϊκό Κόμμα, από το, μέχρι το 2027 ε, ε, υποτίθεται εξασφαλίζει τη ροή και τον όγκο νερού στον τάγο. Δηλαδή μας λέει και λέει σε εσά ότι μέχρι το 2027 ε, θα είναι δεδομένη η κανονική ροή του ποταμιού. Ναι, άμα του, του παίρνεις όμως το καθερό νερό, είναι πολύ δύσκολο να είναι σε καλή κατάσταση το ποτάμι. πριν από δύο χρόνια είχαμε έρθει ξανά στην Επιτροπή σας και ζητήσαμε βοήθεια. Και επειδή στην Ισπανία μας γράφουν κανονικά, για να το πω έτσι, και τους ενδιαφέρει περισσότερο να πηγαίνει το νερό στο Λεβάντε, στην Ανατολική Ισπανία, γιατί εκεί έχουν περισσότερους ψήφους και το ιστορικό είναι άρεο κατοικημένο. Επειδή λοιπόν δεν ξέρουμε σε ποιον απευθυνθούμε, ερχόμαστε σε εσά, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα παράπονά μας. Και κοιτάξτε, αυτές οι φωτογραφίες δεν είναι το 60 ή το 70, είναι σημερινές φωτογραφίες και δεν είναι επεισοδιακές ή περιστασιακές. Είναι ένα ποτάμι που φεύγει στα 400 χιλιόμετρα μέσα από αυτούς τους σωλήνες γίνεται η εκτροπή για να πάνε να ποτίζουν εντατικές καλλιέργειες. Και εμείς αυτό που θέλουμε είναι να ξαναβρούμε το ποτάμι μας, αυτή την κήτη που βλέπετε που το χάσαμε με την εκτροπή και με την αύξηση των λιμάτων. Αυτό θέλουμε να αλλάξει και ζητάμε από εσάς δράση. Και βεβαίως να δώστε συνέχεια σε αυτή την αναφορά και στα παράπονα και τις καταγγελίες που έχουμε κάνει με πάρα πολύ μεγάλη τεκμηρίωση κάπου να πάνε. Γιατί η κυβέρνηση της Ισπανίας σας εμπέζει, δεν σας λέει την αλήθεια και δεν πρόκειται να οδηγηθεί πουθενά με το νέο σχέδιο που έχει καταθέσει. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. And... Ευχαριστούμε πολύ. Λάβαμε από την Κομισιόν πολύ λεπτομερή περιγραφή και απάντηση για όλα όσα έχει κάνει μέχρι τώρα και θα δώσω γι' αυτό το λόγο στον εκπρόσωπό της, στην Λούρδα Αρβαρέγιος, στην εκπρόσωπό της. Ευχαριστώ πολύ. Όντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει την καταγγελία σας. Ανοίξαμε μια ανταλλαγή ε, πληροφοριών με τις αρχές της Ισπανίας. Από το 2014 αρχές του έτους έγιναν διάφορες αλληλογραφίες. Με τελευταία αυτή του Δεκεμβρίου τώρα έχουμε όλα τα στοιχεία στη διάθεσή μας, τα αξιολογούμε αν υπάρχουν ε, ενδείξεις ότι παραβιάζεται η κοινοτική νομοθεσία, ιδιαίτερα η οδηγία για τα ύδατα και για τα πτηνά. Από την άλλη, σε ό,τι αφορά το υδρολογικό σχέδιο, τα έχουμε ξαναπεί αυτά ε, το Δεκέμβριο εδώ στην Επιτροπή σας μετά από την καθυστερημένη έγκριση του υδρολογικού σχεδίου, που μέχρι τον Απρίλιο του 2014 δεν είχε εγκριθεί, η ε, αξιολόγηση της Επιτροπής τώρα ολοκληρώνεται και η έκθεσή της θα ε, δημοσιευτεί το Μάρτιο, ελπίζουμε, αυτό είναι ο στόχος μας. Το θέμα τώρα, ε, το να υπάρχει αρκετός όγκος και αρκετή ποιότητα νερού, για να είναι εξασφαλισμένη η καλή υδρολογική κατάσταση των υδάτων, και η διατήρηση των προστατευμένων περιοχών είναι προτεραιότητα, όπως καταλαβαίνετε, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το βλέπουμε σε μεγάλο βάθος και σας έχω πει και πάλι στο παρελθόν ότι στην αξιολόγηση κάναμε μια διμερή συνάντηση το Νοέμβριο με τις αρμόδιες Ισπανικές Αρχές και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι σε βάθος ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Η έκθεση αξιολόγηση, παραλαμβάνω, θα δημοσιευθεί το Μάρτιο. Λυπούμε, αλλά δεν μπορώ να ε, επεκταθώ σε περισσότερε λεπτομέρειε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μα από το 2012 έχουμε εμεί αυτή την αναφορά και η πιο πρόσφατη απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι του Ιουλίου 2014 και προφανώς αξιολογείται ακόμα τα πράγματα. Νομίζω ότι μας εξηγήσατε παρκώς αυτή τη στιγμή για ποιο λόγο δεν είχαμε περαιτέρω πληροφορίες από το Δεκέμβριο και μετά. κύριος Γκουτιέρες έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Εμείς, οι σοσιαλιστές, υποστηρίζουμε την αναφορά αυτή από πλευρά των ε, αναφερμένων και εγώ κατάγομαι από την Εσκαλώνα που βρέχεται από το ποταμό Αλμπέρτσε που είναι παραπόταμος του Τάγου και γνωρίζω πολύ καλά σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα ποτάμια αυτά η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα αυτή τη στιγμή παραβιάζεται. Γιατί δεν υπάρχει επαρκή ρούς ούτε σε όγκο ούτε σε ποιότητα προφανώς όταν είναι τόσο λίγο το νερό που τρέχει στην κήτη. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ε, αυτή η αναφορά ε, βρίσκει πολύ μεγάλη κοινωνική απήχηση. Η πλατφόρμα ε, αυτή ε, βρίσκει στο πλευρό της τους Δήμους, συντριπτική πλειοψηφία, το λαό, την κοινωνία, τους πολιτικούς φορείς και ζητούν να υπάρχει επαρκής ροή στο ποτάμι. Μια ελάχιστη ποσότητα και ένας όγκος για το περιβάλλον και για την οικολογική αηφορία και του Τάχου και του Αλμπέρτσε, του Τάγου συγγνώμη, για ε, να υπάρξει επαρκής ποσότητα ε, χωρίς αυτή να εκτρέπεται προς άλλη γεωγραφική περιοχή. Είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό. Δεν υπάρχει σε άλλο κράτος μέλος αυτό που συμβαίνει. Ε, το νέο υδρολογικό σχέδιο που έχει εγκριθεί και που τώρα αξιολογείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τα αυτά τα δύο. Ούτε τον αρκετό όγκο και τη ροή για να διατηρείται το ποτάμι, ούτε την ποιότητα των υδάτων. Θα πρέπει λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά, λένε οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες. Ας ελπίσουμε να δούμε την έκθεση το Μάρτιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το υδρολογικό σχέδιο της Λεκάνης του Τάγου και να δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα και πώς παραβιάζεται, γιατί παραβιάζεται η νομοθεσία. Και είναι μεγάλο πολιτικό πρόβλημα και μέγας ο περιβαλλοντικός κίνδυνος που θα πρέπει εμείς από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να καταδείξουμε και να αποκρούσουμε. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι η ομάδα των σοσιαλιστών και δημοκρατών υποστηρίζει το να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να λυθούν αυτά τα σοβαρά προβλήματα. Δεν είναι μόνο περιβαλλοντικά, είναι και κοινωνικά και οικονομικά. Thank you for your contribution. Σας ευχαριστούμε. Να σας πω ότι εμείς καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια να μην δώσουμε πολιτικό χαρακτήρα στις αναφορές. Είμαστε Επιτροπή Αναφορών και κάθε πολιτική ομάδα είναι εξίσου υπεύθυνη για να ακούει τους αναφέροντες και για να καταλήγει σε κάποια συμπεράσματα. Είναι σημαντικό λοιπόν να μην πολιτικοποιούμε τις αναφορές γιατί τελικά ζημιώνουμε την αξία τους, ζημιώνουμε την ισχύ τους, αν κάνουμε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ θλιβερές αυτές οι φωτογραφίες που βλέπουμε. Τόσο αφρό, τόσα νεκρά ψάρια μέσα στο ποτάμι. Το 70 αυτό το βλέπαμε σε όλα τα ευρωπαϊκά ποτάμια. Τέτοιες εικόνες είναι γνωστές. Κανονικά αυτά θα έπρεπε να ανήκουν στο παρελθόν. Θα έπρεπε να είχαμε διδαχτεί από την καταστροφή αυτή. Στην απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγώ τη βλέπω. Ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, λέτε ότι παραβιάζεται ο νόμος. Μετά στη δεύτερη απάντησή σας λέτε ότι α, θα το μελετήσουμε, θα το εξτάσουμε, θα το αξιολογήσουμε κτλ. Το είπε και η πρόεδρος προηγουμένως. Πολλέ αναφορές από την Ισπανία έχουμε και θα πρέπει να προβληματιστούμε. Για ποιο λόγο, γιατί τόσες ισπανικές αναφορές εδώ. Και ξέρω ότι δεν φτάνουν και όλες. Υπάρχουν πολλές πλατφόρμες, πολλές ενώσει, πολλή δουλειά που γίνεται και δεν φτάνει μέχρι εδώ. Με διάφορους οργανισμούς, ενώσεις, κατοίκων και γειτόνων που δεν φτάνουν ποτέ στην Επιτροπή μα. Κατά τη γνώμη μου, δεν σέβονται οι αρχές την κοινοτική νομοθεσία, ούτε καν τη δική τους, την εθνική. Και αυτό είναι επιδημία, δεν είναι ένα απλό σύμπτωμα από εδώ και από εκεί περιστασιακά. Είναι κάτι ευρύτερο στην Ισπανία και θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να κάνει κάτι πολύ σημαντικό εδώ, να το κοιτάξει τι τρέχει στην Ισπανία. Α, και όχι μόνο στην Ισπανία, κατά τα άλλα υπάρχουν και άλλες χώρες φυσικά που δεν τηρούν την νομοθεσία. Αλλά με τόσες πολλές αναφορές και τόσες πολλές περιπτώσεις υπάρχει μια πολύ μεγάλη περίπτωση στην Ισπανία που θέλει ε, γιατριά. Η κυρία Αλμπιόλ. Τι τρέχει στο βασίλειο της Ισπανίας. Θα ήταν πολύ ε, δύσκολο να το συζητήσουμε εδώ και και πολύ χρόνο. Πρέπει να δούμε τι τρέχει με τα ποτάμια στην Ισπανία. Στην Ισπανία το νερό έχει μπει στην υπηρεσία ιδιωτικών συμφερόντων. Έχει μπει ε, και στην υπηρεσία διαφόρων οικιστικών συμφερόντων και διαφόρων πάρκων ε, θεματικών και εμπορικών συμφερόντων. Αυτό το έχει βάλει η κυβέρνηση υπεράνω της ζωής και των ποταμών μας. Το βλέπουμε και στον Τάγο ποταμό, αλλά και σε άλλα πολλά ακόμα ποτάμια. Εμείς τι θέλουμε να υπάρξει επαρκής ροή για να παραμείνει ζωντανό το ποτάμι αυτό. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Και αυτό συνάδει με όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Λοιπόν, αυτή η, οδηγία, η αναφορά συγγνώμη, θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Πριν από λίγες εβδομάδες είδαμε για τον Εύρο ποταμό, τον Ισπανικό Έμπρο, ε, μια αντίστοιχη περίπτωση και αναφορά. θα μπορούσαμε να κάνουμε μια αποστολή εκεί, μια αντιπροσωπεία να στείλουμε για να δούμε επιτόπου πώς έχει η κατάσταση και του τάγου. Προφανώς και θέλουμε να παραμείνει ανοιχτή οδηγία. Γιατί είπε και εκπρόσωπος της Επιτροπής ότι μέχρι το Μάρτιο δεν θα έχει έρθει η έκθεση της Κομισιόν. Ελπίζω μέχρι το Μάρτιο, μη τι άλλο, να παραμείνει ανοιχτή αναφορά και έχει σημασία να γίνει και επιτόπου επίσκεψη για να δούμε με τα μάτια μας περί πρόκειται. Ευχαριστώ. Mm, ναι, Ρώσα, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω ε, τους αναφέροντες που ήρθαν εδώ. Η Ισπανία μετά τη Γερμανία είναι η δεύτερη χώρα που ε, έχει τις περισσότερες αναφορές. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν λειτουργούν καλά οι Ισπανικές αρχές. Μήπως επειδή ξέρουν το δρόμο οι Ισπανοί πολίτες, ξέρουν τις διαδικασίες, έχουμε φέρει το Κοινοβούλιο κοντά στους πολίτες, γι' αυτό και έρχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι πολίτες που διαμαρτύρονται, καταγγέλουν κτλ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πάει κάτι στραβά στην Ισπανία, γιατί για το ναι. περιβάλλον, είτε... γιατί μην πολιτικοποιείτε εδώ πέρα ε, την Επιτροπή. Εμείς δεν έχουμε αυτό το ρόλο. Καταργείται ο ρόλος μας αν το πολιτικοποιούμε. Βεβαίως η αναφορά θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή μέχρι να γνωρίσουμε τι φρονεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι λέει για το υδρολογικό σχέδιο και τις ε, λεκάνες απορροής. Επ' ευκαιρία να σας πω ότι ούτε ο κύριος Κανιέτη ούτε καμία άλλη αρχή ξυπνάει μια ωραία μέρα και λέει τι να κάνω σήμερα να πάω να καταστρέψω τον τάγο ή κανένα άλλο ποτάμι. Δεν το κάνει από καπρίτσιο. Υπάρχουν Υπουργεία και το Υπουργείο Γεωργίας και νόμοι και οδηγίες και τα πάντα. Έχει κάνει υδρολογικά σχέδια η κυβέρνηση, αυτά αξιολογούνται τώρα και στον Έμπρο το ίδιο είχαμε πει. Το Μάρτιο θα φέρει την ανάλυση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιστέψτε με, όλες οι δημοκρατικές κυβερνήσεις αυτού του κόσμου τηρούν τους, κόσμ, τους νόμους. Και η Ισπανική κυβέρνηση, ακόμα και αν δεν σας αρέσει αυτό. Ε, ωραία, να μην είναι ανοιχτή αναφορά. Αν τηρείται ο νόμος ε, θαυμάσια, αν δεν τηρείται να διορθωθεί. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι σκόπι μου ούτε καλή ιδέα να χειραγωγείται αυτή την Επιτροπή μας για σκοπούς πολιτικούς. Ευχαριστώ. Κύριε Σεμπαστιά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Το μόνο που θέλω εγώ να κάνω είναι να βάλω μια απόχρωση εδώ. Η δική μου συμμαχία που εκπροσωπώ ε, περιλαμβάνει και το κόμμα της ε, Καστήλης, γιατί ε, είναι μια περιοχή Καστήλη που πλήττεται πάρα πολύ και ενδιαφέρεται να αποκατασταθεί το ποτάμι. Και έχουμε και το κόμμα Κομπρομής που είναι από την αυτόνομη περιφέρεια της Βαλένθια, που δεν μου αρέσει η όρος Λεβάντε, η Ανατολή που χρησιμοποίησαν οι αναφέροντες. Δεν πρόκειται ε, εδώ για ένα αγώνα, μια αντιπαλότητα μεταξύ των διαφόρων περιφερειών. Είναι τι χρήση θέλουμε να δίνουμε στα νερά των ποταμών μας. Ε, είναι μια μάχη συμφερόντων, γιατί παίρνουν το νερό από το ποτάμι και θέλουν να πάνε να ποτίζουν εκεί τις καλλιέργειε. Ε, θα πρέπει λοιπόν πρώτα να σεβαστούμε την ε, κήτη του ποταμού, τη ροή που χρειάζεται για να μην ε, ξεραθεί και από εκεί και πέρα βλέπουμε αν θα έχουμε βιομηχανική χρήση, γεωργική χρήση και πού θα πηγαίνει και ποιες καλλιέργειες θα ποτίζει. Θα κάνουμε τα βήματα με τη σειρά ένα-ένα γιατί αν χάσουμε την περιβαλλοντική λογική θα χάσουμε και το ποτάμι. Και δεν χρειάζονται αυτές οι αντιπαλότητες μεταξύ των περιφερειών. Ελπίζουμε να βρεθεί μια καλή λύση και καλύτερη για το ποτάμι. Λοιπόν, απόλυτα συνετικά αυτή τη φορά αποφασίζουμε να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτήν και να ευχαριστήσουμε όμως εν προκειμένου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το κάνουμε αυτό πολύ συχνά. Πρέπει όμως να πούμε ότι εν προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια. Ξεκίνησαν διαδικασίες επί παραβάση. Αυτή τη στιγμή δίνουν συνέχεια σε αυτές τις διαδικασίες. Έλαβαν δηλαδή τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι Ισπανικές αρχές θα συμμορφωθούν με την απόφαση του 10 και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει τις δικαστικές διαδικασίες που ξεκίνησε. Επίσης γνωρίζουμε πλέον ότι το Μάρτιο θα κοινοποιηθεί η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα έχουμε δηλαδή την πλήρη αυτή αξιολόγηση. Συνεπώς σας προτείνω να θέσουμε εκ νέου την αφορά αυτή για τη συνεδρίαση που θα κάνουμε τον Μάιο. Μέχρι τότε θα έχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Και κατά αυτόν τον τρόπο ασκούμε πίεση όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει το εξαιρετικό της έργο, αλλά ασκούμε πίεση και σε όλους τους συναδέλφους και ιδίως στους Ισπανούς συναδέλφους να συνεχίσουν να διερευνούν εξονυχιστικά όλα σαν συμβαίνουν στην περιοχή του ποταμού Τάγου. Συμφωνούμε? Πολύ ωραία. Και ξέρετε, φτάσαμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Σας ευχαριστώ όλους για την συμμετοχή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήσασταν σύντομοι στις παρεμβάσεις σας. Ήσασταν πάρα πολύ αποτελεσματικοί. Θα σας δω αύριο και στις 5.30 θα ξεκινήσει η συνεδρίαση των συντονιστών. Σύντομο διάλειμμα για καφέ λοιπόν.